Υπενθυμίζω ότι αύριο την 5η Πρωτη μαρτιου πρόκειται να προβούμε στην εκλογή νέου αντιπρόεδρου του, του Κοινοβουλίου συνδέα του κ. Τσανέσκη και έχουμε δύο υποψηφιότητε. Πρώτα-πρώτα του κ. Σδίσλαβ Κράσνοντέμψκη, κατά πρόταση τη ομάδα ECR και του Ιντρικ Ταρά από το, το βουλευτέ οι οποίοι πληρούν το ελάχιστο απαιτούμενο. Ε, Επίση, ε, ε, διορίστηκε ο κύριο Στάκουλα ω μέλο του ηλεκτρικού Συνεδρίου, οπότε χειρεύει έδρα την 1η του 2018. Mr. Ο κύριο Στάκουλα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είναι η τελευταία μου ημέρα ως Ευρωβουλευτή. Από αύριο αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου στο ελεκτικό συνέδριο στο Λουξεμβούργο. Υπηρέτησα στο θεσμικό αυτό όργανο ως ε, μέλος για 13 πολύ απολαυστικά έτη και τα επόμενα 6 χρόνια θα μου δημιουργήσουν ε, ε, νέες προκλήσεις και μάλιστα έχω και κάποια νοσταλγία για τα χρόνια που αφήνω πίσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και εσάς και τους προκατόχους σας τους συναδέλφους μου ευρωβουλευτές και το ικανό και με πολλά προσόντα προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τάκουλα. Οι καλύτερες ευχές μας σας συνοδεύουν για τα νέα σας ε, καθήκοντα. Ε, οπωσδήποτε και θα συνεχίσουμε να έχουμε επαφή θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τον προπολογισμό της Ένωσης. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Οι αρμόδιες